Dear colleagues, let's uh, move to the uh, agenda item number 16, which is the briefing on the parliament. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Ε, το οποίο αφορά την ενημέρωση για τις εκλογές που έγιναν στο Κοσμοπέδιο στις 6 Οκτωβρίου. Είχαμε προώρες εκλογές τον Οκτώβριο όπως σας είπα η αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον κύριο Αντρέι Κόβατσεφ ε, και ήταν κομμάτι της ε, αποστολής παρατήρησης εκλογών ε, υπό την ηγεσία της κυρίας Βιόλα Φων Καραμόν Τομπαντέλ η οποία είναι βουλευτής της Επιτροπής μας και είναι μόνιμη ησυχήτρια για το Κοσμοπέδιο. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία αυτών των εκλογών. Ελπίζουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσει τις σχετικές μεταρρυθμίσεις ε, προς όφελος όλων των πολιτών του Κοσμοπεδίου και της περιοχής. Ελπίζουμε επίσης ότι οι αρχές ε, θα αναστείλουν τους δασμούς που επιβλήθηκαν στην Σερβία και τη Βοσνία Ριζεκοβίνη για να επανέλθουν στον διάλογο με το Βελιγράδι. Τώρα θα δώσω τον λόγο του συναδέλφους μας που ήταν τμήμα της αποστολής παρατήρησης των εκλογών. Την κυρία Βιόλα Φων Κραμών. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο. Μια που η ενημέρωση συνήθως είναι κάτι το τεχνικό να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις ε. σε σχέση με το Στις προηγούμενες μέρες είχαμε κάποια θετικά μηνύματα είχαμε κάποιες ε, πολύ θετικές αντιμετωπίσεις είχαμε μια πλήρη αποστολή Είχαμε 18 μακροχρόνιους παρατηρητές, 36 βράχοι πρόθεσμους και μαζί με τους συναδέλφους είχαμε 108 παρατηρητές συνολικά. Και μας υποδέχτηκαν θερμά στο Κοσφοπέδιο οι Κοσοβαροί, Αλβανοί, Σέρβοι και και βεβαίως ε, θα έλεγα ότι είναι μία από τις ε, καλύτερες ε, εκλογές που έχουμε παρακολουθήσει από ό,τι μου και οι άλλοι Θα έλεγα λοιπόν ότι είχαμε μια πάρα πολύ θετική αξιολόγηση, μια πολύ καλή συνεργασία με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Λάβαμε μια απόφαση στις 9 Σεπτεμβρίου ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έλαβε μια διοικητική οδηγία ότι μόνο κοσοβάρικα χαρτιά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, κάτι το οποίο αμφισβήτησε η Σεύσκα λίστα, γιατί αποτελούσε ζήτημα από ό,τι φαίνεται, ειδικά για τους εκπροσώπους της Σέρψκα λίστα, αλλά τελικά την ημέρα των εκλογών δεν προκάλεσε προβλήματα και οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είδαν απτές αποδείξεις για το ότι ο κόσμος δεν είχε την δυνατότητα να εκδώσει καινούργια ταυτότητα. Οπότε υποθέτουμε ότι όλα πήγαν καλά. Σε γενικέ γραμμές ήταν ανταγωνιστικές οι εκλογές, υπήρξε ελεύθερη ε, προεκλογική εκστρατεία. Στις ε, σερβικές ε, περιοχές υπήρχε όμως εκφοβισμός των υποψηφίων που δεν ήταν τη ΣΕΠΣΚΑ λίστα η οποία κατήφθηνε τους Σέρβους να ψηφίσουν μόνο αυτό το κόμμα, ενώ έλεγαν ότι οι αντίπαλοι ήταν αντισέρβοι. Ένα πρόβλημα οπωσδήποτε το οποίο ανέφεραν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ε, και βεβαίω αυτό αφορά δικαιώματα του συνέρχεστε των εκλογών και Θεωρούμε άρα ότι οι σερβικές περιοχές ε, δεν ε, ήταν ιδανικές οι εκλογές. Η ελευθερία των ΜΜΕ έγινε σεβαστή. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ε, με μια συνολική κάλυψη και διάφορες προεκλογικές συζητήσεις. Το νομικό πλαίσιο παραμένει το ίδιο όπως τις προηγούμενες εκλογές. Δεν ήδη ε, έχουν βρεθεί κάποια ζητήματα τα οποία θα ρυθμιστούν όπως παραδείγματο χάνει το ότι προκυρήθηκαν πολύ σύντομα οι εκλογές και ότι ε, διάφορα ζητήματα αριθμίζονται μόνο από δευτερογενή νομοθεσία. Επίσης ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα, σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ στην εκστρατεία αυτή από πολιτικά κόμματα και η έλλειψη διαφάνειας παραμένει ένα μεγάλο ζήτημα. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η ακρίβεια και αξιοπιστία των εκλογικών καταλόγων. Τελικοί εκλογικοί κατάλογοι περιέχουν 1,1 εκατομμύρια ψηφοφόρους, δηλαδή περισσότεροι ψηφοφόροι από τον πληθυσμό λόγω του μεγάλου αριθμού ε, διασποράς ε, αλλά και θανόντων εν τω μεταξύ. Επίσης ε, θετικό ήταν ότι η προσέλευση ήταν πολύ μεγαλύτερη, 10% περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Έφτασε το 44% και αυτά για την ώρα μπορώ να δώσω τον λόγο στην ε, συνάδελφο επικεφαλής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Έχω πολύ λεπτομερείς πληροφορίες ε, τεχνικές, ε, δεν ξέρω καλύτερα να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Κόβατσεφ, να πω ότι έχουμε έναν προσκεκλημένο σήμερα. Έχουμε τον κύριο Νίκα εδώ πέρα, πρεσβευτή του Κοσφοπεδίου. Καλώ ήρθατε. Θα κύριο Κόβατσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε για την εξαιρετική σα ε, δουλειά ω παρατηρητή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και συμφωνώ με τα συμπεράσματα που μόλι περιγράψατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του συναδέλφου μου που συμμετείχαν στην αποστολή Εκλογική παρατηρήση στο Κωσυφοπέδιο, Μάντελ, Φραντ. Ιντσερ Φραντ Σαντώνε. Ευχαριστούμε, δείξατε μεγάλη αφοσίωση. Να σας πω τώρα τις παρατηρήσεις μας τον περασμένο μήνα. Οι εκλογές άλλαξαν τα πράγματα στο Παίδιο Για πρώτη φορά μετά από την ε, ανεξαρτησία η πλειοψηφία στο Παίδιο υποστήριξε την αντιπολέτευση. Η κυβέρνηση αναγνώρισε την ήττα της ε, η έκβαση των εκλογών είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα στο κοσυφοπαίδιο για την παγίωση της δημοκρατίας. Οι εκλογές στο κοσυφοπαίδιο γενικά ε, έτυχαν καλή διαχείριση και ανταγωνισμού ε, σε όλη την εκστρατεία, σε όλη τη χώρα, αλλά παρατηρήσαμε, όπως αναφέρθηκε ήδη, και ήταν αναμενόμενο κάποια προβλήματα, όπως είπε η κυρία Φωνκραμών, στην περιοχή των ε, Κωσοβάρων Σέρβων, όχι μόνο στο Βόρα, όπου τα διεθνή πρότυπα δεν ε, τηρήθηκαν στην εκλογική διαδικασία. Και η Σέρψκα λίστα προσπαθεί να μονοπολίσει ε, ε προσπαθεί να μονοπολίσει την ψηφό των Σέρβων ε, του Κωσυφοπεδίου. Για τις αρχές του Κωσόβου έχουν αφοσιωθεί για να συνεχιστεί η επιδίωξη τη δημοκρατία χρειάζεται περισσότερη συνοχή για την αντιμετώπιση συστηματικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν σε παλιότερε αποστολέ και που ακόμα δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα σημεία που ανέφερα εγώ και στην Πρίστινα. Ένα σημαντικό θέμα είναι τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο δεν εγγυάται τη διαφάνεια και την ακαιρεότητα όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες των κομμάτων. Πολλά πολιτικά κόμματα ερμηνεύουν τον νόμο ως ότι απαιτείται να αναφέρουν τι ε, δαπάνε μόνο κατά την προεκλογική εκστρατεία, που αυτή τη στιγμή ήταν πολύ σύντομη σε αυτή την περίπτωση. Αυτό μειώνει σημαντικά τη διαφάνεια. Επιπροσθέτω, έχουμε ακούσει ισχυρισμού ότι το κυβερνών κόμμα έχει εκχωρήσει ε, δημοσίε συμβάσει σε μεγάλου δωρετέ. Ε, αυτό είναι γόνιμο έδαφο για τη διαφθορά. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρατήρησε τα εξή τη διαδικασίες μέχρι σήμερα. Ήταν θετική εμπειρία, είμαστε ικανοποιημένοι με τις εκλογές, έγιναν μετάξι και ηρεμά χωρίς σημαντικά περιστατικά. Υπήρξαν κάποιε παρατυπίε στις διαδικασίες, αλλά περιορισμένε. Συγχαίρω την εκπροσώπηση των μελών εθνικών μειονοτήτων μεταξύ των οποίων και Ρωμά σε ορισμένους ε, σε ορισμένα εκλογικά ε, τμήματα που επισκεφθήκαμε η εκπροσώπηση των γυναικών είναι ένα βασικό ζήτημα για το μέλλον της ε, δημοκρατίας στο Κωσυφοπαίδιο. ο κάποιες θετικές εξελίξεις, ειδικότερα ε, που το 30% των υποψηφίων ε, ως ποσόστοση επιτεύχθη. Αλλά παρατηρούμε ότι οι πλατφόρμες ε, των πολιτικών κομμάτων δεν ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα των φύλων. Συμπερασματικά θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντική η σταθερότητα για το πεδίο. Οι εκλογές του 2019 ήταν τελευταία σε μια σειρά ε, πρόωρων ε, εκλογών ε, κοινοβουλευτικών στο πεδίο. Αυτό δεν προωθεί τη σταθερότητα θα δημιουργηθεί τώρα το νέο κοινοβούλιο και ελπίζω η επιστοποίηση των αποτελεσμάτων να μην ε, χρειαστεί πολύ καιρό. Χρειάζεται το κοσυφοπαίδιο μια νέα κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον. Μια νέα κυβέρνηση που θα μπορέσει να ενισχύσει το κράτο δικαίου και να υλοποιήσει τι ε, θεμελιώδει που απαιτούνται στο κοσυφοπαίδιο και για το λαό του. Υπάρχουν πολλέ ακόμα λεπτομέρειε, αλλά όπω είπε η κυρία Φωνκραμών, προτιμώ να γίνει συζήτηση εδώ στην ΑΦΕΤ για κάποιε λεπτομέρειε, αν χρειαστεί. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σε αυτό το ζήτημα. Thank you, sir. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να μιλήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και εγώ με την παρουσίαση των συναδέλφων και από την ε, επικεφαλής κυρία Βονκραμών. Και εγώ συμμετείχα στην αποστολή. Ήθελα και εγώ να τονίσω ότι και εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές ήταν ε, πολύ καλά οργανωμένες, με κάποιες δυσκολίες φυσικά που δεν οφείλονται μόνο σε αυτά που επισημάναμε, λόγω του ότι ήταν γρήγορες και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Αυτές οι ξαφνικέ εκλογές δεν δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να υπάρξει επαρκής οργάνωση με τρόπο που ενδεχομένω θα ήταν δυνατό ε, εάν ε, είχαν προγραμματιστεί, ε, αν δεν ήταν πρόορες αυτές οι εκλογές. Ε, υπήρξαν κάποιες δυσκολίες. Κάτι που θέλω να προσθέσω που ήταν πολύ θετικό ήταν ε, η συμμετοχή τόσων πολλών νέων ανθρώπων. Και όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν στις εκλογές. Αυτό είναι καλό σημάδι για το μέλλον, αν μη τι άλλο, της χώρας. Ε, δεδομένου ότι δείχνει αυτό ότι υπάρχει ελπίδα, ελπίδα για αλλαγή ε, θετική. Και ήθελα επίσης να συμφωνήσω και με αυτά που υπόθηκαν για το ζήτημα των φίλων. Πιστεύω ότι και αυτό είναι σημαντικό εγχείρημα το οποίο πρέπει να μην ξεχνάμε όχι μόνο με ποσοστώσεις, δεν φτάνουν οι ποσοστώσεις, οι πρέπει να αντιμετωπιστεί και με πολιτικές. Οπότε γενικά ήταν εξαιρετική η αποστολή. Εγώ ίδια πήγα στο Μητρόβιτσα, στο βόρεια πλευρά. Εκεί ήταν κάπως ε, πιο πολλωμένες οι εκλογές. Και ελπίζω ότι θα έχουμε και καλύτερες εξελίξεις όσον αφορά την κατάσταση στις χώρες όσον αφορά την Αλβανία και τους ε, κατοίκους του Κωσυφοπεδίου που, που είναι στους έργους του Κωσυφοπεδίου. Αυτά από πλευράς μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντσί για τα σχόλιά σας και την άποψή σας και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μάνδελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι κύριε Πρέσβη, συμφωνώ με όλα όσα αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους που πήγαν σε αυτή την ωραία χώρα, την νεότερη χώρα της Ευρώπης με την ευκαιρία των εκλογών. Να μην επαναλάβω ότι προελέχθη. Αλλά θέλω να εστιάσουμε προσοχή μας στο εξή που είναι σημαντικό για μένα, για τις μελλοντικές εκλογές, την στάση των ε, κομμάτων που ζήτησαν να οριστούν μέλη Επιτροπής στις εκλογικές επιτροπές σε όλα τα κέντρα, σε όλη τη χώρα σε σχέση με την υποχρέωση ορισμού τέτοιων ε, ε, μελών των επιτροπών στα εκλογικά κέντρα και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκλογικοί αντιπρόσωποι σε συγκεκριμένη περιοχή όρισαν ε, εκπροσώπους και πολλές φορές είχαμε τα κόμματα των μειονοτήτων, εθνικών μειονοτήτων, δεν όρισαν εκλογικό αντιπρόσωπο. Οπότε, είναι ενιαία η χώρα, όλοι είναι πολίτες του Κωσόβου, έχουν αυτό το τόσο σύγχρονο σύνταγμα που κατοχυρώνει δικαιώματα μειονοτήτων και στη Βουλή Άρα θα πρέπει να είναι σαφές ότι θα πρέπει όλα τα κόμματα να ορίζουν εκλογικού αντιπροσώπους. Ακόμα και εκεί που δεν έχουν πολλού οπαδού, πολλά μέλη. Ήταν επομένω ομαδική δουλειά. Και έτσι οδηγούμεθα σε περισσότερη αλληλοκατανόηση στη χώρα μεταξύ όλων των εθνοτικών ομάδων, γιατί υποχρεωτικά εξορισμού συνεργάζονται στα εκλογικά κέντρα. Άρα, αυτή είναι η σύσταση προς τα πολιτικά κόμματα για μέλους της εκλογής να ορίζουν εκλογικούς αντιπρόσωπους. Ήθελα να πω κάτι για την ισότητα ανδρών και γυναικών, την ισομέρη, ισομερή τέλο πάντων εκπροσώπηση, τα είπαμε. Αλλά η γενική ε, εντύπωση είναι ότι όλα πήγαν καλά. Ήταν πολύ καλά οργανωμένε αυτέ οι εκλογέ. Ευχαριστώ κύριε Μάντελ. Έτερο. thank you very much. Um, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ εργάζομαι στην ε, αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη χώρα αυτή και έχω παραστεί ως παρατηρήτρια σε προηγούμενες εκλογές. Είναι σημαντικό, θεωρώ, να υπάρχει συνέχεια. Σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα στο παρελθόν, τι κλίμα επικρατεί. Ε, όχι, δεν μην έχουμε κάθε μέρα εκλογέ όμως. Υπάρχει αίσθηση ότι η χώρα πρόδευε. Και εμείς βέβαια στη Βρετανία έχουμε τις εκλογές που η μία διδέχεται την άλλη και αυτό μπορεί να είναι προσταθεροποιητικό, αλλά πολλές φορές αυτό μπορεί να δίνει δυναμισμό στον κόσμο. Και ιδίως στις καινούργιες ευάλωτες δημοκρατίες. Εμείς εκφράζουμε τη φιλία μας, τη συμπαραστασή μας στο κοσυφοπαίδιο και αυτό έχει σχέση με το πώς φερόμεθα ως παρατηρητές εκλογές. Για μένα όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Πρέπει να συνεχίσουμε να συμπαριστάμεθα στην χώρα. Από κάθε θέση και ως παρατηρητές της εκλογές. Έτσι θα συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τη χώρα. Ευχαριστούμε κύριε Γουόρντ. Ήταν ο τελευταίο συνάδελφο που έχει ζητήσει το λόγο. Οπότε τελειώσαμε και αυτό σήμερα σήμερα σε διάταξη και έχω κάποιες ανακοινώσεις Οι τακτικές μας συνεδριάσεις ως ΑΦΕΤ ε, θα γίνουν στις 18 11 3 η ώρα. Στη συνέχεια, 25 Νοεμβρίου, Στρασβούργο, ή 7. Αλλά πριν από αυτέ τι τακτέ συνεδριάσει θα έχουμε και μια έκτακτη συνάντηση άφετη και ντέλα στις 11 Νοεμβρίου, Δευτέρα. Θα έχουμε ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό του Σουδάν. Επαναλαμβάνω. 11 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Πέρα στη συνεδρία σου. Ευχαριστώ.